Θα δώσω το λόγο στον κύριο Πρωθυπουργό Βίκτορα Ορμπάν, εξ του Συμβουλίου. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχετε τον λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε Μπαρόσο, κυρίες και κύριοι βουλευτέ. Σήμερα θα σας κάνω μία σύντομη επισκόπηση της Ουγγρικής Προεδρίας. Είμαστε ικανοποιημένοι γιατί πριν από έξι μήνες είχατε την καλοσύνη να με καλέσετε πάλι εδώ στην Ολομέλεια και σας είχα παρουσιάσει το πρόγραμμα της Ουγγρικής Προεδρίας. Είχαμε σε αυτό αναφέρει τους στόχους μας και μετά από έξι μήνες είναι εύκολο να κάνει κανείς μια σύγκριση μεταξύ των προγραμματικών δηλώσεων και των επιτευγμάτων της Προεδρίας. Αφού θέλουμε να κάνουμε την αξιολόγηση θα μπορούσαμε να πούμε ότι πετύχαμε απολύτως όλους μας τους στόχους όπως τους είχαμε καθορίσει τότε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την προηγούμενη από εμά Βελγική Προεδρία που έκανε πολύ καλή προπαρασκευαστική δουλειά για μας καθώς και στον πρόεδρο Χέρζη Μπούζεκ γιατί τον Ιανουάριο ήδη είχα πει ότι θέλαμε η Προεδρία μας να είναι φιλική προς το Κοινοβούλιο. Γιατί για διάλογο χρειάζονται δύο και η συνεργασία είναι, με το Κοινοβούλιο είναι κάτι που για μας υπήρξε πολύ ενδιαφέρον και χρήσιμο. Γι' αυτό ευχαριστώ τον κύριο Μπούζεκ, αλλά τώρα ευχαριστώ και τον κύριο Μπαρόσο, διότι για να επιτύχει μια Προεδρία πρέπει το Συμβούλιο να κάνει τεράστιες προσπάθειες και ευχαριστώ τον κύριο Μπαρόσο γιατί και στα πιο δύσκολα θέματα ήταν πολύ ανοιχτός και ειλικρινής και στα επαγγελματικά και στα ανθρώπινα. Επίσης ευχαριστώ τέλος το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σύνολό του αλλά και τον κύριο Ντόλ ιδιαίτερα και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος η Προεδρία πάντοτε διαχωρίζει μεν τη δουλειά της από εσωτερικά πολιτικά θέματα, αλλά αυτό δεν πραγματοποιείται ποτέ και γι' αυτό πρέπει πάντοτε, χρειάζεται πάντοτε η Προεδρία να έχει κάποια πολιτική στήριξη και ο κύριος Ντόλμας τη χορήγησε και μας το κατέστη δυνατόν, μας κατέστησε δυνατόν να εργαστούμε ήρεμα και αποτελεσματικά. Θέλαμε η Ευρώπη να ενδυναμωθεί περισσότερο από ό,τι πριν από έξι μήνες και έγινε αυτό. Όταν πριν από 13 χρόνια για πρώτη φορά ως Πρωθυπουργό συνεργάστηκα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θυμάμαι ότι οι συναντήσεις εκείνες έγιναν με πνεύμα οραματικότητας και αισιοδοξία με μεγάλη ορμή και ενεργητικότητα. Πριν λοιπόν από αυτά τα 13 χρόνια ακόμη γινόταν η προσπάθεια της επανένωσης, της δημιουργίας της ενιαίας αγοράς και του ενιαίου νομίσματος. Και τότε φαινόταν πιθανόν το 2020 να είμαστε η πιο ανεπτυγμένη περιφέρεια της Ένωσης. Δεν φαινόταν ακατόρθωτο. Επίσης θυμάμαι ότι εμείς οι Ούγγροι τότε δεν υποφέραμε από καμία κρίση, ούτε είχαμε αμφιβολίες και ευρωσκεπτικισμό, προσβλέπαμε στο μέλλον με μεγάλη αισιοδοξία. Γι' αυτό κυρίες και κύριοι, Κάνοντας αυτήν τη σύντομη αποκόπηση θα ήθελα να πω ότι σήμερα κατ' εμένα η Ευρωπαϊκή Ένωση πράγματι έχει ενδυναμωθεί περισσότερο από ό,τι πριν από έξι μήνες. Είναι δυνατότερη τώρα παρά το ότι υπέστη τρεις πληγές κατάστηθα την κρίση της Ευρωζώνης, την πυρηνική τραγωδία στην Ιαπωνία και τις προκλήσεις από τις αλλαγές στη Βόρεια Αφρική. Και οι τρεις αυτές εξελίξεις απέτησαν ανταπόκριση από την Ένωση η οποία κατάφερε να ανταποκριθεί όντως στις προκλήσεις αυτές χωρίς να χρειαστεί να μετατρέψει, να μεταποιήσει το εξαμηνιαίο μας πρόγραμμα. Ενδυναμώθηκε λοιπόν η Ευρώπη σε σύγκριση με πριν από έξι μήνες. Αν και δεν το δέχονται αυτό όλοι. Εμείς εδώ προσπαθούμε στην Ένωση να διασφαλίσουμε ότι οι πολίτες παρά την ελληνική κρίση και την εμβάθυνση της γενικότερης κρίσης στα δημοσιονομικά, μπορούν να στηριχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα, τις θεμελιώδεις της αρχές. Γιατί αν δεν μπορέσουμε να πετύχουμε, να έχουμε μία επιτυχή ανταπόκριση στην ελληνική κρίση, τότε δυστυχώς θα ήταν μάταιο να λέμε ότι ενδυναμώθηκε η Ένωση. Μόνο αν μπορέσουμε να έχουμε μία συγκεκριμένη απάντηση στην κρίση αυτή θα μπορέσουμε να πούμε ότι πετύχαμε. Κυρίες και κύριοι λοιπόν, επαναλαμβάνω ότι η Ευρώπη δυναμώθηκε σε σύγκριση με πριν από 6 μήνες διότι κατάφερε να αποτρέψει, να δημιουργήσει τους μηχανισμούς αποτροπής τέτοιων κρίσεων που δεν υπήρχαν πριν από 6 μήνες. Παραδείγματο χάρη το ευρωπαϊκό εξάμεινο που έδειξε στους πολίτες της Ευρώπης ότι τώρα υπάρχουν τα εργαλεία που μπορούν να αποτρέψουν κρίσεις του ενιαίου νομίσματος. Το ίδιο θα μπορούσα να πω και για τα περίφημα 6 μέτρα το 6 pack. που ελπίζουμε να, εγκριθεί, να εγκριθούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τα εργαλεία για να ανταποκριθούμε και να αποτρέψουμε κρίσεις. Αυτές οι αποφάσεις λοιπόν λήφθησαν το τελευταίο εξάμεινο αλλά και για έναν άλλο λόγο μπορούμε να πούμε ότι ενδυναμώθηκε η Ευρώπη γιατί τώρα έχουμε μια στρατηγική που επίσης δεν υπήρχε προηγουμένως και η οποία δεν έχει σημασία μόνο ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά και δίνει την ευκαιρία να διασφαλίσουμε ότι τα εκατομμύρια των Ευρωπαίων πολιτών θα έχουν δικαίωμα πλήρους συμπερίληψής τους στην ε, αγορά εργασίας. Και αυτό δεν αφορά μόνο την κοινότητα των Ρώμα, είναι μια γενικότερη ενδυνάμωση της Ευρώπης. Που μιλώ για το δεύτερο μακροοικονομικό πρόγραμμα ανάπτυξης των περιφερειών με τη στρατηγική του Δουνάβεως η οποία συμπεριλαμβάνει 8 χώρες μέλη και 6 άλλες χώρες. εάν εγκριθεί τελικά που είναι μεγάλη η πιθανότητα να εγκριθεί, τότε θα μπορούμε να πούμε ότι υπήρξε ακόμη, είναι και αυτό ένα επίτευγμα. Η Ευρώπη λοιπόν είναι ισχυρότερη από ό,τι πριν από έξι μήνες διότι η Ουγγρική Προεδρία κατέληξε και τις διαπραγματεύσεις, τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Κροατία. Αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα αυτή, αλλά δίνει νέες προοπτικές και για άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων τους δίνει νέες προοπτικές. Εδώ λοιπόν μπορούμε να πούμε συνοπτικά ότι πρόκειται πάλι για επιτυχία. Υπήρξε ένα μνημόνιο για τη διεύρυνση προς τα Δυτικά Βαλκάνια γενικότερα. Άλλος λόγος ενδυνάμωσης της Ένωσης αυτή τη στιγμή μπορούμε να προστατεύσουμε τα σύνορά μας αποτελεσματικότερα από ό,τι πριν από έξι μήνες γιατί ελήφθησαν αποφάσεις που μας δίνουν τη δυνατότητα να προστατεύσουμε τα εξωτερικά μας σύνορα κατά παρανόμων μεταναστευτικών ροών. Πρόκειται λοιπόν για εμβάθυνση και διεύρυνση των λειτουργιών της Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να σας θυμίσω ότι υπάρχει και κάτι άλλο που ανέλαβε η Προεδρία μας που είναι η διαθεσμική συνεργασία για την αποτροπή διαφωνιών και συγκρούσεων. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έχει διεκπαιρεώσει δεκάδες θέματα με επιτυχή συνεργασία και καταλήξαμε σε συμφωνία ως προς το πώς πρέπει το Κοινοβούλιο να συμπεριλαμβάνεται στην προετοιμασία των πολιετών δημοσιονομικών προοπτικών. Και εγώ προσωπικά ανέλαβα εδώ προσπάθειες και συνεννοήσεις με τον πρόεδρο Βαν Ρόμπαϊ και τον πρόεδρο Μπαρόσο. Εννέα φορές συνάντησα τον πρόεδρο Μπούσεκ Στόχος λοιπόν όλων αυτών των συναντήσεων ήταν να διασφαλιστεί η διαθεσμική συνεργασία ως το δυνατόν πιο απρόσκοπτα. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μου επισκέφθηκα όλους τους Πρωθυπουργούς της Ένωσης ώστε να λαμβάνονται πιο επικοδομητικά οι κοινέ αποφάσεις. Ελπίζουμε η επόμενη Πολωνική Προεδρία να συνεχίσει να προστατεύει, να προωθεί την καλή φήμη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης και νομίζω ότι την προετοιμάσαμε πολύ σωστά και εμείς. Το γενικότερο συμπέρασμά μου λοιπόν είναι ότι ίσως η Ουγγρική Προεδρία και οπωσδήποτε η Πολωνική θα σας πείσουν ότι η απόφαση που ελήφθη για τη διεύρυνση προς τις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης ήταν σοφή απόφαση γιατί έδωσε στην Ένωση μεγαλύτερη ορμή και ζωτικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρωθυπουργέ για την παρέμβαση αυτή. Όπως ε, ξέρουμε η Ουγγρική Προεδρία είχε να αντιμετωπίσει άπειρα προβλήματα, δηλαδή ανέκυψε εν μέσω κρίσης και θα πρέπει να εξευρεθεί ένας τρόπος για να ανταποκριθεί η Ουγγρική Προεδρία σε αυτούς τους μεγάλους κινδύνους και στην κρίση αυτή. Γι' αυτό ακούσαμε με μεγάλη προσοχή όλα όσα μας είπατε. Τώρα θα γίνει συζήτηση επί του θέματος και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το μνημόνιο που μου αποστήλατε και καθώς και στους άλλους και στους πρωθυπουργούς και την καγκελάριο των κρατών μελών. Πρόκειται για ένα μνημόνιο το οποίο σχετίζεται με τα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να τονίσω ότι ο Πρωθυπουργό Όρμπαν μίλησε για τα Δυτικά Βαλκάνια και την επανένωση της Ευρώπης, η οποία έλαβε χώρα το 2004 και τώρα θα πρέπει να συμπληρώσουμε την διαδικασία επανένωσης. Επίσης αναφέρθηκε στην κατάσταση στις μεμονωμένες χώρες και μίλησε για ένα στρατηγικό πρόγραμμα το οποίο θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Θα ήθελα να πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάντα υποστήριζε τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα Δυτικά Βαλκάνια. Μετά βεβαίως την τήρηση των κριτηρίων, διότι αυτό αποτελεί απαράβατο όρο για τη διεύρυνση. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζωζέ Μανουέλ Μπαρόζο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, διακεκριμένα μέλη της Ουγγρικής Κυβέρνησης, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι. Αντιμέτωποι με πολύ δύσκολες συνθήκες, η Ουγγαρία ανταποκρίθηκε με πολύ ικανή Προεδρία του Συμβουλίου. Γενικότερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί καλύτερα να αντιμετωπίσει ευκαιρίες και δυσκολίες. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Όρμπαν και όλοι, όλους τους συνεργάτες του για την αφοσίωση στη δουλειά. Κατά την Ουγγρική Προεδρία στο Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση επέτυχε το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο, ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με την Κροατία, ε, υποστήριξε την Αραβική Άνοιξη, προχώρησε στην στρατηγική των Ρώμα. Χάραξε νέες στρατηγικές, καλά αποτελέσματα όλα αυτά. Θέλω επίσης να τονίσω τον ανοιχτό διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια του δημοσιονομικού πλαισίου. Τον περασμένο Νοέμβριο άρχισε ένας δομημένος διάλογος. Ε, αυτό συνέπεσε με την Ουγγρική Προεδρία. Ο πρόεδρος Μπούζεκ, ο πρωθυπουργός Όρμπαν και εγώ συναντηθήκαμε επανειλημμένα για να ανταλλάξουμε απόψεις πριν από την υιοθέτηση των προτάσεων της Κομισιόν που έχετε Πρόκειται για ρεαλιστικό και φιλόδοξο προϋπολογισμό και για την επένδυση στην μελλοντική μεγέθυνση. Αυτή η πρακτική των διαβουλεύσεων ε, των διοργανικών μεταξύ των θεσμικών οργάνων τώρα έχει παγιωθεί και ο Πρωθυπουργό Τούσκ μου επιβεβαίωσε ότι η Πολωνική Προεδρία θα ακολουθήσει προς την ίδια κατεύθυνση. Άρχισε ο διάλογος, θα συνεχιστεί και θα δώσει καρπούς. Εξετάζουμε την κρίση για να χαράξουμε πολιτική. Χρειαζόμαστε εργαλεία για να επανέλθει σε τροχιά, να παραμείνει σε τροχιά η Ευρώπη και αυτό δεν είναι μικρό επίτευγμα. Μια εποχή όπου ε, αλλάζουν διεθνώς πολλά πράγματα, εμείς επιλέξαμε να επιμείνουμε στην αλληλεπίδραση θεμάτων οικονομίας ε, και θεμάτων όπως μετανάστευση. Ε, η οικονομία. Η μεγέθυνση ήταν μεγάλη προτεραιότητα στην Ουγγρική Προεδρία και θα παραμείνει και στην Πολωνική. Στο οικονομικό κλίμα σήμερα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. 1,8% ε, αναμένεται ως ανάπτυξη για το 2011 και η ανεργία είναι απαράδεκτα υψηλή, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων. Οι αποκλήσει ε, μεταξύ κρατών μελών εξακολουθούν να είναι υπερβολικές και χώρες ε, όπως η Ελλάδα περπατούν, σχηνοβατούν. Ε, αυτό που διακυβεύεται είναι το μέλλον της κοινωνικής οικονομίας της αγοράς ή ο ρόλος μας ως Ευρώπη στον κόσμο. Η Κομισιόν λοιπόν θέλει να υποβάλει σημαντικέ προτάσεις για την οικονομική διακυβέρνηση μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ των συνομοθετών τελική ε, συμφωνία του πακέτου για την οικονομική διακυβέρνηση διαφαίνεται τώρα και θα ήθελα τα δύο θεσμικά, άλλα θεσμικά όργανα να επισπεύσουν και να ανταποκριθούν στο σημαντικό πακέτο το οποίο στηρίζεται στην εξαιρετική δουλειά που έκανε ο εισηγητής. Από τη δική μας την πλευρά η Κομισιόν θα συνεχίσει να εργάζεται σκληρά για να δώσει αποτελέσματα σημαντικά σε τομείς σημαντικούς ε, ε, πράξη για την ενιαία αγορά. για παράδειγμα, μέχρι το τέλος του χρόνου θέλουμε να ολοκληρωθούν οι προτάσεις, ελπίζοντας ότι θα εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2012 από Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Χαίρομαι γιατί βλέπω πρώιμους καρπούς ε, ιδιαίτερα σε θέματα όπου προτάθηκαν μεταρρυθμίσεις ε, και ε, συμφωνήθηκαν και δύο κανονισμοί για τη βελτιωμένη συνεργασία, ούτω ώστε να έχουμε σε θέματα διανοητικής ε, ιδιοκτησίας ευρωπαϊκή πατέντα. Ε, είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε για να ε, μειωθεί το κόστος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη κατά 80% και θα καλύπτονται 25 κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να έχουμε φιλικές ε, καινοτομίε και έχουν και μεγάλη οικονομική αξία. Θα τερματίσουμε την απαράδεκτη κατάσταση όπου η απόκτηση μιας πατέντας είναι δεκαπλάσια σε αξία στην Ευρώπη από ό,τι στις είπα. Η ευρωπαϊκή δράση μπορεί λοιπόν να συμπληρώσει τις ευρωπαϊκές δράσεις για την ανταγωνιστικότητα. Κάτι άλλο σημαντικό κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αφορά στη μετανάστευση, η οποία είναι ένα θέμα συναισθηματικά φορτισμένο. Σήμερα αντιμετωπίζει δυσκολίες και προκλήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, μετά τα ε, γεγονότα της περαμεσμένης άνοιξης. Ως Ένωση όμως δράσαμε για να προασπίσουμε την ασφάλεια και την ελευθερία. Ε, συμφωνήθηκε ο νέος κανονισμός ε, για τη Frontex πριν από δύο εβδομάδες. Μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις στα πλαίσια της διακυβέρνησης του Σέγγεν και τις εθνικές δράσεις που ε, θα υπονομεύσουν ενδεχομένω βασικές αρχές μας όπως η ελεύθερη διακίνηση προσώπων και τον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο χωρίς σύνορα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα υποβάλλει συγκεκριμένε προτάσεις ε, για παρακολούθηση σε ευρωπαϊκή βάση. Λίγο πιο αργά διακόπτει ο πρόεδρος Μπούζεκα γιατί οι διερμηνείς δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν. Ε, σας παρακαλώ να διαβάζετε λίγο αργότερα. Έλεγα λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα θα υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για ευρωπαϊκή βάση παρακολούθηση και σύστημα αξιολόγησης βέβαια που θα συμπληρώνεται από έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό ε, για το άσυλο συμφωνήσαμε ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε το κοινό σύστημα ασύλου μέχρι το 2012. Οι προτάσεις της Κομισιόν ήδη βρίσκονται επιτάπητος και έχω εμπιστοσύνη ότι έχουμε τη δυναμική που χρειάζεται για να ολοκληρώσουμε το σκοπό αυτό. Χαίρομαι γιατί η Ουγγρική Προεδρία έκανε μεγάλο βήμα μπροστά για τους Ρωμά το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις στρατηγικές ενσωμάτες των Ρωμά εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα μας βοηθήσει να σταματήσουμε σε τέσσερις τομείς την απομόνωση, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία, ε, και άλλες, ε, άλλους τομείς ε, ήταν πραγματικά πολύ ευαίσθητος ο χειρισμός αυτής της συμφωνίας. Τώρα, για την προσχώρηση της Κροατίας, η πρόοδη. Οι διαβουλεύσεις ολοκληρώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και θα υπογράφει η συμφωνία προσχώρησης μέχρι το τέλος αυτού του έτους. Κατά τη γνώμη της Κομισιόν, η Κροατία θα μπορούσε να γίνει το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 1η Ιουλίου 2013. Είμαστε αυστηροί αλλά δικαίοι και θα συνεχίσουμε να είμαστε μέχρι την ώρα της προσχώρησης. Πιστεύω ότι θα ενισχυθεί η ευρωπαϊκή οικογένεια έτσι, αλλά θα ε, προωθηθεί και η συμφιλίωση και η σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα ήθελα να αποτίσω φορό τιμή ε, στην στεναρά υποστήριξη που είχαμε κατά την καθοδήγηση αυτή της διαδικασίας που έδωσε πρακτικό νόημα στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής. Χαιρετίζω την ε, υποστήριξη της ε, Ουγγαρίας ε, στο θέμα αυτό του μέλλοντος των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης, ορίσαμε τη νέα στρατηγική βοήθεια για σύνδεση, ανάπτυξη σε εταιρική σχέση με εξηγήτονες. Ο συνολικός στόχος είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής για τα 150 εκατομμύρια ανθρώπων που ζουν στην περιοχή. Φέτος επίσης ήταν σημαντική χρονιά για την πολιτική γειτονίας η πολιτική γειτονία περισσότερο από ποτέ βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ένωσης. Αντιμετωπίσαμε προβλήματα των νοτίων γειτόνων. Όχι μόνο υποστηρίξαμε πολιτικά την Αραβική Άνοιξη, αλλά και επιτόπου με ανθρωπιστικά μέτρα και δράσεις ε, και ορίσαμε μια στρατηγική για τη δημοκρατία και την ε, ευημερία. Θα ήθελα τέλος να πω, αγαπητά μέλη, ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στην επένδυση στο μέλλον. Η Ουγγρική Προεδρία ανταποκρίθηκε και η στενή συνεργασία με τη νέα Πολωνική Προεδρία θα εξυπηρετήσει καλά την Ένωση. Θα διασφαλίσει τη συνέχεια στο έργο του Συμβουλίου και θα επιτρέψει επικοδομητικές ανταλλαγές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μπορέσαμε να προχωρήσουμε την Ευρωπαϊκή Ατζέντα αυτό το εξάμεινο και είμαι βέβαιος ότι το επόμενο εξάμεινο θα μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω στα επιτεύγματα για να έχουμε σημαντικές ε, επιτυχίες για την Ένωσή μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ τον ε, κύριο Πρόεδρο Μπαρόζο εξ ονόματος ε, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ε, ο πρόεδρος Ζεφ Ντόλ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνέδελφοι, η Ουγγρική Προεδρία κατέδειξε ότι η εκπεριτροπής Προεδρία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα θεσμικά μας ζητήματα. Είχε να αντιμετωπίσει πολλά μέτωπα η συγκεκριμένη Προεδρία ε, την επιτυχία του πρώτου ευρωπαϊκού εξαμήνου, την κρίση και θέματα κοινωνικής συνοχής μέσα στα πλαίσια της ΚΑΠ, της διατροφικής ασφάλειας, της εσωτερικής αγοράς και της στρατηγικής στην περιοχή του Δούναβη, καθώς και της, την πολιτική ενέργειας. Εξωτερικό μέτωπο για τη διεύρυνση προς την Κροατία και συνεννόηση με τους λαούς της Μεσογείου και με τους φίλους μας, τους Ιάπωνες. Αγαπητέ κύριε Ορμπάν, θα ήθελα να σας πω, να σας ευχαριστήσω καταρχήν και ιδιαίτερα την Ένι ε, Κόγκερη, την ε, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, η οποία βοήθησε ιδιαίτερα για την κατάληξη θεμάτων όπως η Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και η Κοινοτική Μέθοδος. Επίσης, καταφέραμε να επιτύχουμε τους στόχους μας κατά 85-90% και νομίζω ότι, αγαπητοί συνάδελφοι, χωρίς οικονομική διακυβέρνηση δεν θα υπάρχει σταθερό ευρώ και χωρίς σταθερό ευρώ δεν θα μπορέσουμε να κερδίσουμε στον τομέα της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής, η οποία θα είναι σχεδόν μηδενική. Αυτή είναι η πεποίθηση του ΕΛΚ. Θα ήθελα να τονίσω ότι από τον Ιανουάριο επιτελέστη μεγάλη πρόοδος στις κοινέ πολιτικές όπως την πολιτική συνοχής με τη Συμφωνία του Φεβρουαρίου είτε πρόκειται για την ΚΑΠ με την ε, συμφωνία του Μαρτίου για μία μεταρρύθμιση, λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση των τιμών ε, πρώτων υλών και τροφίμων είτε πρόκειται για την ενέργεια και την καινοτομία, όπου ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με το θέμα το Φεβρουάριο για ένα ολόκληρο μήνα μετά από την τραγωδία της Φουκουσίμα. Επίσης, μιλήσαμε για την ε, εσωτερική αγορά με την ε, συμφωνία επί του Single Market Act. Μιλάμε για μία δύσκολη πολιτικο-οικονομική συγκυρία. Επίσης φτάσαμε σε μια συγκεκριμένη πολιτική υπέρ των Ρωμά, όπου εσείς κύριε Ορμπάν συμφιλιώσατε τους Ευρωπαίους επί του θέματος και σας ευχαριστώ όλος ιδιαιτέρως για αυτό. Επίσης είχαμε μεγάλες επιτυχίες στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων. Μίλησα για την πρόοδο στην περίπτωση της Κροατίας και οι 27 έδωσαν συμφώνησαν έτσι ώστε να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις από τον Ιανουάριο. Αυτή η διεύρυνση είναι πολύ καλή και για τους Κροάτες αλλά και για τα Βαλκάνια που θα βασίζονται σε μία απτή ευρωπαϊκή πολιτική. Επίσης, τα θέματα της Μεσογείου σας απασχόλησαν. Η Ευρώπη κατέδειξε την αλληλεγγύη της και στα λόγια αλλά και στις πράξεις και μπόρεσε να επιλύσει τα θέματα μετανάστευσης, ιδιαίτερα στα Ιταλικά ε, παράλια, στις Ιταλικές ακτές και μίλησε υπέρ μιας πολιτικής μετανάστευσης. Επίσης προσχώρησαν στο χώρο Σέγγεν η Βουλγαρία και η Ρουμανία γιατί τηρούν πράγματι τους κανόνες Καταβλήθηκαν μεγάλες προσπάθειες σε αυτό το τομέα και για άλλη μια φορά ευχαριστούμε ε, την Ουγγρική Προεδρία και ευχόμαστε επιτυχία και για την Πολωνική Προεδρία. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Αντιπρόεδρος Χάνες Βόμποτα έχει το λόγο εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρωθυπουργέ. Δύο καθήκοντα έχει η Προεδρία. Πρέπει να συνεχίσει τους ε, ε, διάφορους φακέλους και να τους ολοκληρώνει τα τρέχοντα και να ασκεί και μια υποδειγματική λειτουργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά το πρώτο θέμα, κύριε Πρωθυπουργέ, θέλω να ευχαριστήσω τους πολιτικούς συνεργάτες σας θερμά, διότι πολλά θέματα ε, λύθηκαν ικανοποιητικά. Ο φάκελος της Κροατίας που με απασχολούσε ιδιαίτερα, η στρατηγική των Ρωμά επίσης. Ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά το δεύτερο θέμα όμως, έχω να κάνω κάποιες κριτικές παρατηρήσεις γιατί και σε ό,τι αφορά το νόμο για τα μέσα ενημέρωσης και το Σύνταγμα, εδώ στο Κοινοβούλιο εκφράσαμε μεγάλη κριτική. Μπορείτε να αντιπαραθέσετε την πρόκειται για εσωτερική πολιτική, αλλά ξέρετε κύριε Πρωθυπουργέ ότι στην Ευρώπη η εσωτερική πολιτική είναι και ευρωπαϊκή πολιτική και αντίστροφα η ευρωπαϊκή πολιτική αντανακλάται και επηρεάζει την εσωτερική. Έτσι λοιπόν είναι θεμητή η ευρωπαϊκή κριτική. Ε, θα έπρεπε να αντιδράσετε παρόλο που ήταν ήπια η κριτική για το νόμο για τα ΜΜΕ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης η Επιτροπή της Βενετίας δεν επέκρινε μόνο τη διαδικασία αλλά και σημαντικά συστατικά στοιχεία ε, της αλλαγής του συντάγματος και ε, άλλοι επίσης σημαίνοντε σημαίνουσες προσωπικότητες έκανα κριτική. Ε, ε είπατε ότι ε, θέλετε να προχωρήσετε το 45. Μεταξύ του 45 και του σήμερα υπάρχει και το 56. Η μεγάλη στόχη, ο πλουραλισμός, η ελευθερία της έκφρασης των μέσων ενημέρωσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να αναφερθεί το έτος 1956 ως το έτος της Μεγάλης Επανάστασης με τις ελευθερίες αυτές ως στόχο που αποτελούν και ευρωπαϊκούς στόχους. Και δεν είναι όπως εσείς τουλάχιστον ως πρόεδρος λέγατε ότι πρόκειται για μια κριτική των σοσιαλιστών προς την κυβέρνησή τους. Είσαστε στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο όταν η Χίλαρη Κλίντον πρόσφατα ε, επέκρινε ε, την πολιτική αυτή ε, και ε, αναφέρθηκε ε, ε, στην ανάγκη για επαγρύπνηση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις. Όλοι πρέπει να επαγρύπνουμε, όχι μόνο στην Ουγγαρία, αλλά λόγω των εξελίξεων αυτών περισσότερο η Ουγγαρία. Έχετε δύο τρίτα πλειοψηφία θεωρητικά, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά σε μια δημοκρατία ευρωπαϊκού τύπου μετράει και η γνώμη των επικριτών, μετράει η γνώμη της αντιπολίτευσης, όχι μόνο αυτά που λέει η πλειοψηφία των δύο τρίτων. Ευχαριστήσατε το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Μόνο το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ευχαριστήσατε. Δικαίωμά σας, παρόλο που ήθιστε ε, οι προεδρίες ε, να μην ευχαριστούν ένα κόμμα μόνο. Αλλά δημοκρατία σημαίνει όχι μόνο, ε, στη δημοκρατία συγκαταλέγονται όχι μόνο οι υποστηρικτές κάποιου αλλά και οι επικριτές. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή δημοκρατία και θα ήθελα να σπαστείτε τους στόχους του πλουραλισμού κάπως περισσότερο. Ε, όπως ε, ε, αναφέρθηκε είναι πολύ σημαντικό οι Ευρωπαίοι να αναλάβουν ευθύνη όλοι και να πούν ναι στον πλουραλισμό, ναι στην ελευθερία έκφρασης, ναι στην ελευθερία της κριτικής που και αυτή συγκαταλέγεται στα δημοκρατικά δικαιώματα ε, ανεξάρτητα από τις πλειοψηφίες ε, που υπάρχουν και οι πολέμοι και οι επικριτές θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Έτσι τουλάχιστον εκλαμβάνουμε εμείς την ουσία της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Κυρία Σβόμποντα, υπάρχει μια μπλε κάρτα για σας. Ο συνάδελφος Πόσελτ. Παρακαλώ, κάντε την ερώτηση. Ναι, κύριε Πρόεδρε, η Ουγγαρία δεν είχε μόνο εξαιρετική προεδρία, αλλά και ένα σύγχρονο δημοκρατικό σύνταγμα. Θα ήθελα να ρωτήσω τον συνάδελφο Σβόμποντα, πιστεύει ότι ο Μπάνκι Μουν, ο οποίος ε, ο, ο Κίμιλ Γιόγκ ο Μπαν Κιμούν θα έπρεπε να ε, ασχολείται ε, περισσότερο ε, με τις δημοκρατικές παραδόσεις των χωρών που εκπροσωπεί στον οργανισμό του ε, ή τι δημοκρατίε. Ο κύριος Μπάνκι Μουν υποστηρίχθηκε στην εκλογή του ως Γενικός Γραμματέας από πολλές δημοκρατίες. Δεύτερον, εγώ ανέφερα πολύ συγκεκριμένα την Επιτροπή της Βενετίας. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν είναι σοσιαλδημοκράτες εκεί, αλλά περισσότερο σχέση έχουν με το δικό σου κόμμα. Η δημοκρατία δεν είναι θέμα κομμάτων είναι θέμα ε, προσωπικής ε, ε, κατανόησης και πολιτικής αυτοκατανόησης. Αυτό ήθελα να τονίσω και προς τον Πρωθυπουργό Ορμπάν. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο Αλεξάνδρ Γκραφ Λάμστορφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, κύριε Πρωθυπουργέ. Η ομάδα μου θεωρεί ότι ήταν δύσκολη η Προεδρία με τη δημοσιονομική κρίση, με τις εξελίξεις στη Φουκουσίμα μας στη Βόρεια Αφρική και κύριε Όρμπαν ε, η κυβέρνησή σας, ο Υπουργός Εξωτερικών σας, ο Υπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, ο κ. Γιώρη ε, πετέλεσαν εξαιρετικό έργο και στην οικονομική πολιτική. Αυτά που επετέφθησαν, τη σταθεροποίηση του ευρώ, σίγουρα πρόκειται για μεγάλη επιτυχία, αλλά παραμένει ένα σημαντικό καθήκον. Η έγκριση του EFSF και η ε, συμφωνία για το ESM είναι σημαντικά επιτεύγματα. Επίσης, το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο, ο συντονισμός τη δημοσιονομική πολιτικής των κρατών είναι πολύ σημαντικό για να αποτρέπεται η συσσόρευση των χρεών που ήταν ε, συνηθισμένο πράγμα κατά το παρελθόν. Κάτι που μένει ανοιχτό είναι το Six Pack, το πακέτο για την οικονομική διακυβέρνηση. Επιμένουμε ως ομάδα και θα συνεχίσουμε να επιμένουμε να έχουμε ενισχυμένο σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης και θα μείνουμε σκληροί και στο θέμα της ειδική πλειοψηφία. Δεν πρέπει να αναβληθεί το θέμα αυτό. Πρέπει να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις. Ο Ζωζεφ Ντόλ είπε ότι ε, είναι πιστικό το πακέτο που ε, θα πρέπει να είναι πιστικό το πακέτο για να υπάρχει σταθερότητα του ευρώ είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί τομεί που είχατε μεγάλη επιτυχία. Η Κροατία αναφέρθηκε, η ολοκλήρωση των ε, ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Συμφωνώ ότι ε, αυτό σημαίνει μεγάλο βήμα για όλη την περιοχή. Βλέπω ε, ο κύριο Σουάμπ, η οδηγία για του καταναλωτέ ολοκληρώθηκε το πλάνο για την απόδοση της ενέργειας επίσης και ένα σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ε, Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας ε, που ανέφερε και ο Πρόεδρος Μπαρόζο και πολλές άλλες επιτυχίες σημείωσε η Προεδρία σας. Κύριε Πρωθυπουργέ, όταν συναντηθήκαμε στη Βουδαπέστη σας είπαμε ότι θα αξιολογήσουμε με δίκαιο τρόπο την Προεδρία σας βλέποντας όμως ε, και Τη εξελίξη στη χώρα σα από τη δική μα σκοπιά, τη φιλελεύθερη. Λυπούμεθα, διότι επισκιάστηκε από τα προβλήματα για τον νόμο για τα ΜΜΕ, θα επιθυμούσαμε ένα άλλο νόμο για τα μέσα ενημέρωση. Η Κομισιόν ε, πέφερε κάποιες ε, τροποποιήσεις, αλλά όχι σε θέματα κλειδιά. Θα θέλαμε επίση η διαδικασία τη επεξεργασία του Συντάγματο να είχε λάβει χώρα σύμφωνα με τι προτάσει τη Επιτροπής της Βενετίας. Νομίζω ότι η επαγρύπνηση των υπόλοιπων Ευρωπαίων για κάθε κράτο μέλο και για το δικό μου θα πρέπει να συνεχιστεί για να συνεχιστεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είτε πρόκειται για την ελευθερία ταξιδίων, για την ελευθερία του τύπου, δεν έχει σημασία. Είναι πολύ σημαντικό. Ε, σύντομα ε, θα επανεισαχθούν τελωνιακοί έλεγχοι στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ θα θέλαμε κάποια πιο στεναρή ε, αντιμετώπιση τα θέματα του Δουβλίνου 2 ε, και η, ελεύθερη, ελευθερία ε, ταξιδίων θα θέλαμε εδώ ε, μεγαλύτερη δέσμευση και από τη δική σας την Προεδρία. Συνολικά μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώσατε μια επιτυχή Προεδρία και θα είμαστε ακόμη πιο χαρούμενοι αν δεν είχαμε αυτές τις εξελίξεις που επεσκίασαν κάποια θετικά, τα θετικά σημεία. Ευχαριστώ, Συμπρόεδρος Κον Μπέντιτ από την ομάδα των Πρασίνων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, πολλές φορές δεν κατανοώ γιατί μιλάμε. Μας είπατε ότι η Ευρώπη είναι δυνατή, μπορεί να δράσει, πρέπει να δράσει. ως μια δύναμη η οποία θα πρέπει να επιβληθεί σε μια δύσκολη πολιτική και οικονομική κατάσταση. Όλοι χειροκροτούν. Μετά διαβάζω. Το 48 δεν δεχτεί δεχτήκαμε τα δόγματα της Βιέννης. Το 90 δεν δεχτήκαμε ή και νωρίτερα δεν δεχτήκαμε το ε, δόγμα της Μόσχας και σήμερα δεν θα δεχτούμε το δόγμα των Βρυξελών. Ποιος το είπε αυτό, ο Βάκλαφ Κλάους, όχι, ο Όρμπαν φέτος και μετά Αναρωτιόμαστε γιατί δεν υπάρχει θετική γνώμη της Ευρώπης στη χώρα τους, διότι υπάρχουν πολιτικοί άνδρες που μιλάνε κατά αυτό τον τρόπο εδώ στις Βρυξέλλες, αλλά διαφορετικά στη χώρα της. Και αυτό αποδυναμώνει την Ευρώπη. Και εσείς είσαστε ένας από αυτούς τους ανθρώπους, κύριε Βικτόρ Ορμπάν, αποδυναμώνετε την Ευρώπη, διότι το πράγμα είναι πάρα πολύ απλό. Εσείς και οι υπάλληλοι σας επιτελέσατε, πολύ καλό έργο. Μιλάμε για μια γενικευμένη σχιζοφρένεια εδώ και για έναν εθνικό κινησμό. Δηλαδή στην η Ουγγαρία τι κάνουμε. Ε, αποδυναμώνουμε αυτό που χτίζουμε στην Ευρώπη. Έχω δίκιο. Έτσι δεν είναι. Δίκιο δεν έχω. Σας ευχαριστώ. θα θέλαμε να ε, ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα στα πλαίσια της νομιμότητας κατά, αυτής, ε, κατά αυτών των διαδηλωτών που θέλουν να προστατεύσουν. Ε, θέλουμε να ε, προστατεύσουμε τα σύνορά μας κατά των έξω δυνάμεων. Τι είχε πει όμως ο Γιάννος Καντάρ, ότι θα πρέπει να επιτελέσουμε το ακριβώς αντίθετο. Αυτό είναι το πρόβλημά σας κύριε Ορμπάν. Δηλαδή το 89 δώσατε ένα μεγάλο αγώνα και στη συνέχεια ήρθατε ε, μη έχοντας εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Είσαστε κατά της δικτατορίας των ε, Βρυξελών. Άρα τι κάνετε ε, στην ουσία δεν έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας. Ίσως έτσι θα καταλαβαίνατε και την ε, θέση της Ευρώπης. Δηλαδή, μιλάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον κύριο Μπαρόζο, ο οποίος ε, μίλησε υπέρ ε, μία συγχώνευσης τύπου, ενώ εσείς δεν το δεχτήκατε. Έχετε ένα ελεύθερο ραδιόφωνο, το Club Radio, το οποίο είναι ελεύθερο. Όλος τυχαίως έρεται η συχνότητα, απαγορεύεται η συχνότητα, ενώ δίνεται αυτή η συχνότητα σε ένα καθολικό ραδιόφωνο. Λέτε ότι είναι κάτι τυχαίο από την ιστορία, όμως δεν ισχύει κάτι τέτοιο μπορείτε να δείχνετε ε, ότι δεν συμφωνείτε, αλλά δεν σας ενδιαφέρει καν, διότι μετά θα προβείτε σε έναν καθαρά εθνικιστικό λόγο, λέγοντας ότι γνωρίζετε τι είναι Ευρώπη. Μιλήσατε υπέρ της ελευθερίας, αλλά δεν σας άκουσα να λέτε πολλά πράγματα υπέρ των διαδηλωτών της Αιγύπτου και της Τινησίας. Στην Κίνα όμως κινείστε πολύ αργά, άρα μην μας λέτε ό,τι θέλετε. Αλλά ως προς το πρόβλημα των συνόρων και τι κάνει η Δανία σήμερα, θα πρέπει η Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πούν ότι αυτή η κατάσταση θα πρέπει να, να σταματήσει Μιλάμε για συμφωνίες ε, Σέγγεν και ούτε η Ουγγαρία ούτε η Δανία μπορούν να εφαρμόσουν μονομερός το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και εάν αλλάξει το ευρωπαϊκό δίκαιο θα αλλάξει με συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και δεν είσαστε στην πλειοψηφία, κύριε Μπαρόζο. Κύριε Ορμπάν, επιτελέσατε καλή εργασία, αλλά εσείς δώσατε μεγάλη μάχη όντας δικτάτορας κατά της δικτατορίας. Ο επόμενος... Ευχαριστώ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο συνάδελφος Ζαχράντιλ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής. Η Ουγγαρία πρέπει να αναγνωριστεί για την εργασία που έχει επιτελέσει κατά την Προεδρία της. Την συγχαίρω ιδιαιτέρως συγχαίρω τη γραμματεία της Προεδρίας που συναντήθηκε μαζί μας πολλές φορές. Πρόκειται για νέα χώρα μέλος και δεν ήταν εύκολο για αυτήν να αναλάβει την Προεδρία αντιμετώπισε και εσωτερικά προβλήματα, τις αλλαγές στη Βόρεια Αφρική και τις προκλήσεις όλες αυτές τις αντιμετώπισε. Η εσωτερική σταθερότητα διατηρήθηκε και τελικά θα ήθελα να εκφράσω και ορισμένες επικρίσεις ή τουλάχιστον ορισμένη τη λύπη μου για ορισμένα πράγματα. Εγώ διαφωνώ με τον κύριο Ορμπάν κάπως, δηλαδή θεωρώ ότι η διεύρυνση προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη δίνει μια νέα δυναμική στην Ευρώπη, αλλά δεν έγινε τελικά αυτό που δηλώνουμε, γιατί οι νέες χώρες γρήγορα συνήθισαν στη γραφειοκρατία και τα τετριμένα που λένε όλοι στην Ευρώπη και δεν άσκησε καμία ιδιαίτερη πολιτική ηγεσία. Θα ήθελα κάποτε ένας πρωθυπουργός στη θέση σας να σηκωθεί και να πει δεν μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια αυτή παπαλαιωμένη πολιτική της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που ίσχυε πριν από 50 χρόνια. Ίσως βέβαια πάλι ο κύριος Κονπεντίτ τότε να τους κατηγορήσει για αντιευρωπαϊστές, αλλά οι πολίτες είμαι σίγουρος ότι θα επικροτήσουν. Ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μίλοσλαβ Ράνσντορφ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ομολογώ ότι εμένα μου αρέσει η Ουγγαρία και ο πολιτισμός της και γι' αυτό ήθελα να δω πώς θα αντιμετώπιζε την προεδρία της. Πρέπει δεν να σας πω ότι απογοητεύτηκα. Πήρα μέρος σε πολλούς τριμερείς διαλόγους, στην τριμερή συνεννόηση με τα τρία όργανα και είδα ότι υπήρχε μια πλήρης έλλειψη προετοιμασίας από την Προεδρία. Συνεχίζοντας αυτά που είπε ο κύριος Ζαχραντήλ θα έλεγα ότι πρόκειται για τη συνέχιση των, της πεπατημένης. Θα μπορούσε κανείς να συνοψίσει την Προεδρία λέγοντας ότι ήταν μηδενική. Για μένα αυτό είναι λυπηρό, ιδιαίτερα λυπηρό, γιατί Επρόκειτο για Προεδρία που αντιμετώπισε προκλήσεις και εσωτερικά και εξωτερικά. Πού εφαρμόστηκε αυτή η ενίσχυση της Ευρώπης που είπε ο κύριος Ορμπάν. Στα μέσα ενημέρωση στην Ουγγαρία, στους Ρωμά, εκεί ναι, εκεί τήρησε στεναρή στάση, καταπιεστική. Κάτε με, το Κοινοβούλιο συγχαίρει υπερβολικά τον εαυτό του. Δεν πρέπει να κάνει μόνο αυτό. Πρέπει κάποτε να βλέπει τα πράγματα και διαφορετικά διότι οι ευκαιρίες που δίνουν οι νέες χώρες μέλη καθώς και οι δικοί μου δεν έχουν τύχη εκμετάλλευσης και στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε ακόμη σημαντικότερες προκλήσεις από ό,τι μέχρι τώρα. Όπως είπε και ο Μέρβιν Μοχάτσκολ πρέπει η αντιμετώπιση να γίνει για να επιβιώσουμε. Ο κ. Είστε από τους λίγους ε, Ευρωπαίους ηγέτες κύριε Ορμπάν που μιλάτε τόσο στεναρά υπέρ της δημοκρατίας και φαντάζομαι ότι δεν θα πτωηθείτε από αυτά που λένε εδώ οι ενωσιοεθνικιστές. Όταν μιλήσατε κατά της δικτατορίας των Βρυξελών και της Μόσχας νομίζω το λέγατε σοβαρά Είστε από τους ηγέτες των ευρωσκεπτικιστών και η εξάμηνη προεδρία σας υπήρξε πράγματι ιστορική διότι τους έξι αυτούς μήνες οι λαοί της Ευρώπης ξύπνησαν επιτέλους και κατάλαβαν ότι είναι τελείως μη δημοκρατικός ο χαρακτήρας της Ένωσης. Αυτό το καταλάβατε μετά τις εκλογές στη Φιλανδία και την καταπληκτική επιτυχία του κόμματος των πραγματικών Φινλανδών καταλάβαμε όλοι ότι δεν θέλουν όλοι οι λαοί να συνεχίσουν με αυτό το αποτυχημένο πρόγραμμα. Και μετά βέβαια υπήρξε και η καταστροφή της Πορτογαλίας και για να επανέλθουμε στην Ελλάδα για το δεύτερο δάνειο Είδαμε τις τρομερές διαδηλώσεις που σημειώθηκαν και εκεί. Αλλά το βασικό στοιχείο της Προεδρίας σας είναι ότι η Δανία στην ουσία έσκησε τη συμφωνία του Σέγγεν. Κατά την εξάμηνη λοιπόν αυτή η Προεδρία έγιναν περισσότερα για να ξυπνήσει η δημοκρατία και το μέλλον του έθνους κράτους από ό,τι προηγουμένως. Και αυτό είναι καλό να το καταλάβουμε έχουν αλλάξει τα πράγματα, έχουμε δει την αρχή του τέλους αυτού του επικίνδυνου ενωσιακού προγράμματος. Σας συγχαίρω κύριε Όρμπαν που το καταλάβατε. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σέγκεντη, μη εγγεγραμμένος. Ναι. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο, αξιότιμα κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη κύριε Πρωθυπουργέ. Επιτρέψτε μου παρακαλώ να εξετάσω δύο θέματα και να κάνω μια ανάλυση της εξάμηνης Ουγγρικής Προεδρίας. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζομαι και αναλύομαι γεγονότα και θα ήθελα να τα αναλύσω μέσα από το Ουγγρικό πρίσμα αντιμετωπίσαμε δύο θέματα. Έχουμε μια οικονομική συμμαχία η οποία δέχεται την κυριαρχία των κρατών εθνών. Αυτή είναι η μία εναλλακτική που δέχεται την κυριαρχία των κρατών και η άλλη ε, προσέγγιση αντιμετωπίζει ως απικίες στα κράτη. Η Ουγγρική Προεδρία ζήτησε να εξετάσουμε τα θέματα αυτά και το θέμα της κυριαρχίας. Το 2004 εκατοντάδες χιλιάδες στην Ουγγαρία ψήφισαν υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί θεωρούσαν ότι οι Ούγγροι στα Καρπάθια θα μπορούσαν να επανενωθούν, να κινούνται ελεύθερα και να νιώσουν μέλη μιας κοινότητας. Α υποθέσουμε ότι η Ουγγρική Προεδρία είναι μια συμβολική Προεδρία και δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια ελιγμών ε, σε εθνικό επίπεδο. Τι γίνεται με το νόμο της ε, σλοβακικής ε, γλώσσας στα διάφορα διατάγματα για τις επιμέρους περιφέρειες. Τι προοπτική έχουν όλα αυτά. Είδαμε ότι δώσατε μάχη για ένα λανθασμένο νόμο για τα μέσα ενημέρωσης. Δεν μας πειράζει η στρατηγική για τους Ρωμά, αλλά μας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν, κατα... καταβάλατε... Ε, δεν μια ουγγρική στρατηγική. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο συνάδελφος Γιώζεφ Σάγερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, λίγες μέρες μετά το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας. Η πρώτη αίσθηση είναι ότι η δουλειά έγινε. Είμαστε περήφανος λαός στην Ουγγαρία ε, και ε, ανταποκρινόμεθα στις υποχρεώσεις που αναλαμβάνουμε. Αυτό έγινε και τώρα. Εμείς ε, μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Λέσχη και ακολουθήσαμε και τηρήσαμε τους κανόνες της. Ο νόμος για τα ΜΜΕ αναφέρθηκε, επικρίσεις ακούστηκαν, ανταποκριθήκαμε και δεν ζητήσαμε καμιά ιδιαίτερη μεταχείριση. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, κυρίες Βόμποντα, θα σας διαβάσω το προήμιο του Ουγγρικού Συντάγματος ε, στα Αγγλικά. Η πρώτη απόφαση είναι η ε, τωρινή μας ε, ελευθερία προήλθε από την ε, Επανάσταση του 1956. Θέλω να πω ότι το Ουγγρικό μας Σύνταγμα σαφώς και αναφέρεται στο 1956 και ε, επί, αυτού ε, στηρίζει τα θεμελία του συντάγματος. Θα ήθελα επίσης ε, να αναφερθώ στην άποψη του κυρίου Κονμπέντιτ που εκφράστηκε ως κοσμοθεωρία σήμερα και είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι βουλευτές εργάστηκαν καλά. Βεβαίως έχουμε και καταγωγής Ρώμα Ευρωβουλευτή Επίσης ε, έχουμε και στεναρούς ηγέτες καταγωγής Ρωμά στη χώρα μου. Ε, ίσως ε, να υπάρχει εδώ μια ε, κρυφή αντίφαση. Εμείς οι Ουγγροί λέμε αυτό που, κάνουμε αυτό που λέμε και υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες το προηγούμενο εξάμεινο για τη στάση μας αυτή. Εδώ βλέπουμε τι θα κάνει το Κοινοβούλιο τις επόμενες ώρες. Υπάρχουν προτάσεις ψηφισμάτων και εξετάζουμε όλο αυτό το θέμα των στεναρών όρων που έχουν ε, τεθεί στα πλαίσια της διαδικασίας τροποποίησης του συντάγματος. Ε, μετά μιλάτε για ε, δικτατορικές πρακτικές. Θα ήθελα επίσης να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο κύριος Όρμπανε όλους τους ευχαρίστησε, όπως και εμείς δεν περιοριστήκαμε σε ένα κόμμα. Ο κύριος ε, Σάμπα Σάντορ Ταμπάτζη. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μπαρόζο, η δήλωσή μου στην αρχή της Ουγγρικής Προεδρίας ισχύει και σήμερα. Είπα ότι κάθε Ούγγρος πατριώτης, είτε πρόκειται από το ΕΛΚ είτε από τους σοσιαλιστές, θα, πρέπει να ασχοληθεί με την υποστήριξη και την επιτυχία της Ουγγρικής Προεδρίας. Οι Ούγγροι διπλωμάτες ε, επιτέλεσαν πολύ καλό έργο για τη διεύρυνση προς την Κροατία και αυτή είναι μια μεγάλη επιτυχία της Προεδρίας. Επίσης, το ε, ε, Ευρωπαϊκό Εξάμεινο καθώς και η πολιτική υπέρ των Ρωμά και του Δούναβη έχουν επιτύχει. Επίσης, προωθήσαμε ένα πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης. Κατά την Προεδρία, οι επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων δεν συναντήθηκαν στην Ουγγαρία, ούτε η Σύνοδος Κορυφής έγινε στην Ουγγαρία. Η εσωτερική πολιτική βεβαίως επισκίασε αυτές τις πολιτικές. Δυστυχώς δεν φτάσαμε σε σωστά αποτελέσματα. Δυστυχώς ο νόμος υπέρ του τύπου, ε, το Σύνταγμα και οι ευρωσκεπτικιστές οδήγησαν σε εξωτερική κατακραυγή. Η Ουγγρική κυβέρνηση απομονώθηκε κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Δυστυχώς επιδεινώθηκε και η κατάσταση ε, προερχόμενη από τις εξωτερικές αντιδράσεις. Καταδικάστηκε ο νόμος για τα μαζικά μέσα ενημέρωσης καταδικάστηκε από την Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τη Γερμανία και άλλες κυβερνήσεις και η γερμανική κυβέρνηση επέκρινε και το Σύνταγμα. Δεν ισχύει το γεγονός ότι η αριστερά της Ευρώπης ε, κατέκρινε την δεξιά της Ουγγαρίας. Δεν θέλουμε να σας ε, δώσουμε μαθήματα δεν θέλουμε να προβαίνουμε να κάνουμε επικρίσεις, να προβαίνουμε σε επικρίσεις, αλλά μας ενδιαφέρει η επιβολή ενός δημοκρατικού συστήματος. Κατά το τελευταίο εξάμεινο η Ουγγρική κυβέρνηση υπέστη πολλές επικρίσεις και οπωσδήποτε δεν είμαστε υπερήφανοι για αυτήν την κατάσταση. Εκ. Δεν πρόκειται μόνο για λήψη αποφάσεων, αλλά οι προεδρίες έχουν και συμβολικό χαρακτήρα, προάγουν ανθρώπινα δικαιώματα, ελευθερία έκφρασης, θεμελιώδεις ε, αξίες. Ε, χαίρομαι λοιπόν γιατί θέσατε επιτάπητο στο ζήτημα των Ρωμά, αλλά λυπούμε διότι εσωτερικά η Ουγγρική κυβέρνηση δεν έδειξε την ίδια δέσμευση σε αυτές τις ε, αρχές εσωτερικά. Ε, η Ουγγρική Προεδρία έκανε πολύ καλή δουλειά διότι επέκτηνε την ευρωπαϊκή οικογένεια για να συμπεριλάβει την Κροατία. με πολύ ικανοποιημένη διότι ολοκληρώθηκαν επί της Προεδρίας σας οι διαπραγματεύσεις γιατί είμαι επικεφαλής της αντιπροσωπείας για την Κροατία. Είναι καλό διότι ε, πετεύχθη ένα ιστορικό, μια ιστορική επιτυχία. Επίσης ε, το φάκελος για την ενέργεια με μεγάλη δεξιοτεχνία προωθήθηκε. Αντιμετωπίστηκαν προβλήματα μετά το υδραγωδία στην ε, Φουκουσίμα, ε, ζητήματα που αφορούν τον ενεργειακό δικό χάρτη. Τέλος κύριε Πρόεδρε, σχετικά με την επόμενη Πολωνική Προεδρία. Ε, για το τελευταίο, μετά το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών για το Περιβάλλον ανησυχώ διότι τα θέματα του κλίματος δεν τα λαμβάνουν τόσο σοβαρά όσο θεωρώ ότι θα έπρεπε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ συνάδελφοι να μιλάτε πιο αργά γιατί οι διερμήνεις μας δεν καταλαβαίνουν, δεν προλαβαίνουν. Dirk Jan Epping. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όποτε έχει προβλήματα η Ένωση αρχίζουν οι ηγέτες της να κατηγορούν τους λεγόμενους λαϊκιστές. Αυτό το κάνει τακτικά ο κύριος Μπαρόσο και ελπίζω να με ακούει τώρα. Αυτό δείχνει ότι απομακρύνονται όλο και περισσότερο από την πραγματικότητα. Οι απλοί άνθρωποι περιμένουν. Τους είπαν ότι θα υπάρξει οικονομική σύγκληση και γίνεται το αντίθετο. Αναρωτιούνται τι θα γίνει ε, με τις οικονομίες μου, με τη σύνταξή μου, ποιο μέλλον θα έχουν τα παιδιά μου. <clears throat> Είναι όλοι αυτοί που αναρωτιούνται αυτά τα πράγματα λαϊκιστές κύριε Μπαρόσο. Το να κατηγορούμε τους άλλους για λαϊκισμό δεν είναι σωστό κύριε Μπαρόσο. Να κοιτάξετε τι κάνετε εσείς. Δίνετε υποσχέσεις που δεν τις εφαρμόζετε. Νομίζω καιρός είναι να αρχίσουμε να ενισχύουμε τα επιτεύγματα της ολοκλήρωσης αντί να χτίζουμε πύργους της Βαβέλ κύριε Μπαρόσο. Δεν είναι τίποτα, δεν υπάρχει τίποτε λαϊκιστικό σε αυτά που λέμε. Αντίθετα τα ευρωομόλογα λένε ότι είναι η λύση για τα χρέη. Πώς μπορούμε να μειώνουμε τα χρέη αντί, ε, κάνοντας, δημιουργώντας ακόμη περισσότερα κύριε Μπαρόζο μου. Η πλειοψηφία εδώ έξω από το κοινοβούλιο αποτελείται από ανθρώπους που αναρωτιούνται Πράγματα για τα οποία δεν έχετε καμία απάντηση κύριε Μπαρόζο μου. Σας ευχαριστώ. Επόμενος μιλητής, ο κύριος Πάσκα που λείπει όμως. Γι' αυτό ο κύριος Λάγκεν. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί πρόεδροι. Νομίζω ότι η Ουγγρική Προεδρία ήταν πολύ επιτυχής, αν λάβουμε υπόψη μας τις προκλήσεις. Αν λάβουμε υπόψη μας την απροθυμία κάποιων κρατών μελών να συμβάλλουν σε κοινή ευρωπαϊκή λύση. Σε ό,τι αφορά την Προεδρία αυτή θα ήθελα να, κάνω, να δώσω συγχαρητήρια. Θέλω να ε, συγχαρώ και την ε, Υπουργό Επιευρωπαϊκών Θεμάτων κυρία Γκέρι. Ε, επίσης ε, θα ήθελα να πω ότι δεν συμφωνώ με τον κύριο Λάμστορφ πώς θα κάνει σωστές προτάσεις μια προεδρία όταν τα μεγάλα κράτη-μέλη συνεχώς μπλοκάρουν τις εξελίξει. Υπάρχουν πολλά σχετικά παραδείγματα. Και εν ώψη των προκλήσεων τα κατάφερε καλά η προεδρία. Αν ε, δούμε την, ε, τις παρεμβάσεις ε, ε ε, Ζαχατήλ, Κονμπέντιτ, Σβόμποντα. Εξαφανίστηκαν όμω, Δεν θέλουν να ακούσουν τι απαντήσει και τα σχόλια επί των δηλώσεών του Είναι άδικο αυτό προ την Ουγγρική Προεδρία. Βεβαίω θα έπρεπε να λύσετε και εσωτερικά προβλήματα. Βεβαίω υπήρξαν και αντιπαραθέσει. Αλλά ε, έχοντα ακούσει τον κύριο Σβόμποντα, ο οποίο δεν επισήλθε στην ουσιαστική ατζέντα της Ουγγρικής ε, Προεδρίας, Πρέπει να πω ότι αυτή ήταν μια, ε, ένας ελιγμός ε, για να μας αποτρέψει από τα σημαντικά θέματα. Βεβαίως δεν μπορούν να λυθούν όλα τα προβλήματα από την Κίνα μέχρι την Νότια Αφρική. Εσείς ε, την Προεδρία σας την ολοκληρώσατε με επιτυχία και αν δούμε ότι εκφράστηκαν ε, και ε, επικρίσεις από τις Βρυξέλλες. Ε, εγώ αυτό θα πρέπει να το δω με κριτικό πνεύμα, διότι ε, οι παρεμβάσεις τους ούτε ήταν πολύ στεναρές, ούτε επέμεινε για αποτελέσματα. Ε, προφανώς η Ουγγρική Προεδρία ήταν σωστή Προεδρία και είχε επιτυχία. Κύριε Λάγκεν, είστε διατεθειμένος να απαντήσετε σε μια ερώτηση με τη μπλε κάρτα, τη διαδικασία της μπλε κάρτας. Ο κύριος Μποστινάρου θέλει να θέσει την ερώτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Λάγκεν, ε, πολύ χαίρομαι που θα σας προκαλέσω. Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο είδατε την ε, γνώμη της Επιτροπής της Βενετίας για το Σύνταγμα της Ουγγαρίας και ποια είναι η γνώμη σας σε σχέση με αυτή την έκθεση η οποία είναι και η πιο επικριτική τα τελευταία 20 χρόνια από ό,τι είδαμε στην Ευρώπη. Ich habe... Ε, Τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας δεν την διάβασα, ούτε διαβάζω ουγγρικά. Διάβασα πολλές αξιολογήσεις που λέγουν ότι το Ουγγρικό Σύνταγμα είναι από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Πολλές φορές ε, ε, κάποιοι ευρωβουλευτές ε, είναι υπερβολικά αυτάρεσκοι και αυτό θα πρέπει να σταματήσει. Ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση αυτή. Η κυρία Τάνια Φαγιώνη. Θα ήθελα να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία για τη μεγάλη της επιτυχία ως προς την προσχώρηση της Κροατίας. Η διαδικασία διεύρυνσης ε, συνεχίζει. Αυτό είναι πολύ θετικό για τα Δυτικά Βαλκάνια και σας συγχαρήκαμε, σας συγχαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό. Αυτό ε, αφορά, τα συγχαρητήριά μας αφορούν και το θέμα των ορομά και τη στρατηγική σας, αλλά μας απασχόλησε το θέμα των εσωτερικών σας θεμάτων, οι εσωτερικές διαφορές σε σχέση με τον νόμο για τα ΜΜΕ και ε, ορίσατε ένα νόμο για, που να αφορά τη δική σας εσωτερική ικανοποίηση. Κύριε Όρμπαν, είσαστε ένα σύμβολο της Ευρώπης. Δεν θα θέλαμε να παλινοδούμε στην Ευρώπη. Αν και η Ουγγρική Προεδρία ε, δεν όρισε κάτι τέτοιο. Ε, ευχόμαστε ότι η Πολωνική Προεδρία θα ε, οδηγήσει, θα οδηγήσει προς την αντίθετη κατεύθυνση. Γκέρενς, Σαρλ Γκέρενς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο πρόεδρος Ορμπάν θεωρεί ότι η Ευρώπη είναι πιο δυνατή σήμερα παρά έξι μήνες πριν. Δεν συμμερίζομαι αυτή σας ε, την παρατήρηση. Η κακοφωνία ήδη από την αρχή της ελληνικής ε, κρίσης δεν ενίσχυσε την Ευρώπη. Η κερδοσκοπία είναι πιο υψηλή από ό,τι έξι μήνες πριν. Η πραγματική Φινλανδοί είναι πιο δυνατή από ό,τι έξι μήνες πριν. Η διεύρυνση δεν θα καταστήσει την Ευρώπη πιο δυνατή παρά μόνο αν διαθέτει κανόνες έτσι ώστε να τηρηθούν τα κριτήρια της Κοπενχάγης από όλα τα κράτη-μέλη. δηλαδή όχι μόνο πριν αλλά και μετά την προσχώρηση των κρατών ως προς τη συμφωνία του χώρου Σέγγεν υπάρχουν πολλοί σκεπτικιστές οι, οι οποίοι έχουν αντιταχθεί σε αυτή τη συμφωνία που είναι πιο δυνατή σήμερα παρά έξι μήνες πριν δυστυχώς. Ο συνάδελφος Πάσκα είναι εδώ και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Βίκτορ Όρμπαν. Αδιαμφισβήτητα η Ουγγρική Προεδρία προσπάθησε να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Και γι' αυτό σας ευχαριστούμε. Η καθημερινή δουλειά αυτού του διοικητικού μηχανισμού όμως επισκιάστηκαν από κάποιες εσωτερικές εξελίξεις στην Ουγγαρία. Γι' αυτό στις Βρυξέλλες ε, συχνά δημιουργήθηκαν παρεξηγήσεις. Ακολούθησε η αναθεωρημένη τροποποίηση που ανέφερε η Επιτροπή της Βενετίας και την ε, έλαβε υπόψη για τη γνωμοδότησή της. Σίγουρα δεν είναι απλό να ικανοποιήσει κανείς όλες τις πλευρές. Ίσως λείπει ακόμη από το Σύνταγμα κάποια κατοχήρωση δικαιωμάτων. Ε, δεν είναι τέλειο το ε, Σύνταγμα. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή, διότι η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων προσπάθησε να ασχοληθεί με αυτά τα ζητήματα μέσα στα πλαίσια και της ΚΟΖΑΚ έτσι ώστε να υπάρχει ευρωπαϊκός προσανατολισμός και της Ουγγρικής Προεδρίας. Η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων θα ήθελα να σας ευχαριστήσει διότι περατώθηκε η έκθεση για την πρωτοβουλία των πολιτών και το, θέμα αυτό προωθήθηκε και από την Υπουργό Γιώρη. Η, η Ουγγαρία μιλάει για μια πιο δυνατή Ευρώπη. Αυτό ήταν το λογότυπό της. Και αυτό θα πρέπει να δούμε κατά πόσο τηρήθηκε. Ε, ζήσατε μία, ένα εξάμεινο χιονοστιβάδων, ε, έναν τυφώνα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι, ε, είναι να δούμε κατά πόσο το σύνταγμά σας, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο το σύνταγμά σας παραβιάζει πτυχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, επειδή είμαι συνταγματολόγος και έχω μελετήσει όλα τα συντάγματα των κρατών μελών, θα πρέπει να πω ότι δεν μπορεί κανείς να παρεμβαίνει στα εσωτερικά θέματα μιας χώρας. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω για την εργασία σας αλλά και για το Σύνταγμα το οποίο ενισχύει τους οικογενειακούς ε, δεσμούς. Η κυρία Έντιτ Χέρτζοκ ε, έχει το λόγο. Αξιότιμα μέλη, ε, δεν ξέρω εάν ε, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ε, αναφέρθηκε πιο πολύ σε εθνικό ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Βρυξέλλες σίγουρα δεν είναι Μόσχα όμως και πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε σεβασμό προς τους ε, ε, ε, υπαλλήλους της Ευρώπης. Πιστεύω λοιπόν ότι ένας από τους αντιπρόεδρους του Κοινοβουλίου είπε κάτι σωστό. Δεν θα μας σταματήσει τίποτε επειδή θα θέλουμε να παραμείνουμε μετριοπαθείς. Η μετριοπάθεια όμως δεν εκφράστηκε στις δικές σας πολιτικές, ιδιαίτερα αν δούμε το δημόσιο τομέα. Η Ουγγαρία είναι σε πόλεμο. Αυτή είναι μια έκφραση που χρησιμοποιήθηκε και αυτή αποσπά... Α, διάκοπη από τον ε, κύριο Μπούζεκ και κυρία Γκουλάρ. Καλημέρα σας κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να βοηθήσω ε, όλες τις ουγγρικές ομάδες με τις οποίες συνεργαστήκαμε. Δεν θα ήθελα όμως να σταθώ σε αυτό. Με εκπλήσει ένα ζήτημα. Ο Ότοφον Φον απεβίωσε κατά το τέλος της Ουγγρικής Προεδρίας και σκέφτομαι τι ήταν η Αυστρο-Ουγγρική Αυτοκρατορία στην αρχή του 20ου αιώνα. Τι θα πρέπει να μας δείξει αυτό, ότι τα κράτη είναι ευάλωτα και όσοι υποδαβλίζουν τον εθνικισμό θα πρέπει να μην ξεχνάνε αυτό το παρελθόν και μην ξεχνάτε ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απεβίωσε ακριβώς γι' αυτό το λόγο, διότι ανβίωσαν εθνικισμοί. Δεν θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει εθνικισμός. Ο κύριος Πρόντι έλεγε πάντα σε, με αυτούς που συγκρίνουν τη δικτατορία των Βρυξελών με την δικτατορία της Μόσχας. Θέλω να μου υπενθυμίσετε πότε προσχωρήσατε στη Σοβιετική Ένωση και όχι στην Ευρωπαϊκή. Η κυρία Βόρτμαν Κόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για τη δέσμευσή της έκανε σημαντική δουλειά για να επιτευχθεί μια συμφωνία για την οικονομική διακυβέρνηση και κατά 98% πραγματοποιήθηκε η συμφωνία αυτή. Κύριε Ουρμπάν, το... ο σκοπός σας ήταν να ενισχυθεί η Ευρώπη. Αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά με μια ισχυρή διακυβερνητική ομάδα και γι' αυτό χαιρετίζω ιδιαίτερα τη δουλειά όλων των συνεργατών και πρεσβευτών. Κατά την αρχή της Προεδρίας σας δηλώσατε ότι θέλατε το Κοινοβούλιο να του φερθείτε σοβαρά και το αποδείξατε αυτό. Γιατί και πολλοί από τους δικούς μας στόχους επετέχθησαν, Δεν μην τους επαναλάβω. Είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο συναποφασίζει επί πολλών σημαντικών θεμάτων. Γι' αυτό τα 2% των εναπομεινών άντων θεμάτων ε, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιτευχθούν και αυτά. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες, προσπάθειες λέγω, ώστε τα 2% που λείπουν να επιτευχθούν και αυτά. Γνωρίζω βέβαια ότι αυτό το 2% που δεν έχει επιτευχθεί υπάρχει, αλλά κάνατε ό,τι μπορούσατε και Χάρη στην προπαρασκευή σας το Σεπτέμβριο νομίζω ότι η επόμενη Προεδρία θα μπορέσει να καταλήξει. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία μου. Ο κύριος Φρεντερίκ Ντάρντεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, απευθύνομαι σε εσά ως μέλος της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων. Έχουν σημειωθεί πρόοδοι σε διάφορα θέματα όπως για τους Ρωμά Αντίθετα όμως από την προηγούμενη Προεδρία που είχε προωθήσει τα κοινωνικά για τους άστεγους, για την καταπολέμηση της ανέχειας, η δική σας Προεδρία λίγα έκανε για τα κοινωνικά. Παρ' όλα αυτά αναφερθήκατε σε θέματα ανάπτυξης και προώθησης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Προτύπου. Δυστυχώς δεν είδαμε τίποτα κατά την εξάμηνη αυτή Προεδρία παρά τις συζητήσει για τα δημοσιονομικά. Δεχτήκατε την κυρίαρχη ιδέα ότι η οικονομική διακυβέρνηση έγκυται κυρίως σε περικοπές στους προϋπολογισμούς, όπως η απόφαση σας, η εσωτερική απόφαση, το Ίδρυμα Πίτλερ, που αναγνωρίζεται διεθνώς και που συμμετέχει στην καταπολέμηση της ανεχίας των παιδών δεν το ενισχύσατε. Δηλαδή δεν κάνατε αυτά που υποσχεθήκατε. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ την Ουγγρική Προεδρία γιατί περισσότερη σημασία έχουν τα επιτεύγματα παρά όσα απέμειναν και θα πρέπει να γίνουν. Είναι γεγονός ότι δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα πρέπει να έχει μακροοικονομικούς στόχους. Ε, δουλειά που έγινε στο θέμα των ρωμά ε, και στα θέματα της ασφάλειας της σέγγεν κτλ. είναι σωστή. αυτό που είναι σημαντικό για να δοθεί συνέχεια είναι να δοθεί έμφαση στην κοινωνική διάσταση που αφορά στην επίτευξη των στόχων 2020 εγώ ε, ως βουλευτής προερχόμενη από την ελλάδα θέλω να ευχαριστήσω την ουγγρική προεδρία για τις προσπάθειες ε, για τη βοήθεια προς τη δημοσιονομική προσαρμογή της χώρας μου και να τονίσω ότι δεν, δεν έχουν σημασία οι ιδιαίτερες διαφορές που υπάρχουν και αυτές είναι στα πλαίσια της δημοκρατίας μέσα στον ελληνικό χώρο. Ε, ως έλληνες αναγνωρίζουμε ότι χωρίς αυτή τη βοήθεια θα είχαμε πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα και άρα αναλαμβάνουμε και τη δέσμευση των υποχρεώσεων και τη συνεργασία και με την εκάστοτε προεδρία και με την ευρωπαϊκή επιτροπή. κύριε πρόεδρε το σημαντικότερο απ' όλα νομίζω είναι ότι πρέπει να υπολογίσουμε πώς μπορεί να επιτευχθούν οι στόχοι 2020 από εδώ και πέρα γιατί λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατευθυντήριες γραμμές της λισαβόνας δεν απέδωσαν αυτό που θέλουμε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you, Madam. The next speaker, Madam Vice President Roberta. Η κυρία Ρομπέρτα Αντζελίλη, αντιπρόεδρος, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, έγινε μεγάλη συζήτηση για το νέο Ουγγρικό Σύνταγμα, αλλά πέρα από τις διαφωνίες θα ήθελα να πω ότι ότι στο σύνταγμα αυτό αναφέρεται το μέλλον των νέων γενεών. Είναι, αναφέρονται οι νέες γενές. Και επειδή υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση για τους νέους και τα παιδιά, φαίνεται ότι η Ουγγρική Προεδρία έδωσε μεγάλη προτεραιότητα στην καταπολέμηση της παιδοπορνογραφίας και της εκμετάλλευσης των ανηλίκων. Εγώ είμαι η συγγήτρια, θα ψηφιστεί η έκθεση αυτή την επόμενη εβδομάδα και πρόκειται για ένα πολύ εύγλωτο μέσο με κυρώσεις υπέρ των θυμάτων της καταπολέμησης του σεξουαλικού τορισμού και της προσέλκυσης των ανηλίκων μέσω διαδικτύου στυλιτεύονται αυτά τα αδικήματα καθώς και η online παιδοπορνογραφία. Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα σημεία που θα ήθελα να υποστηρίξω. Όμως όλα αυτά κατέστησαν δύνατα ακριβώς επειδή υπήρχε μεγάλη ευαισθητοποίηση της Ουγγρικής Προεδρίας επί των θεμάτων αυτών. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκολπέλς έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν ε, δούμε τις απαρχές και ε, την αποδοτικότητά μας, μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες μέτρα σε έναν πολύ ε, σύντομο αγώνα. Δεν ξέρω κατά πόσο λάβαμε υπόψη του στόχος μας, αν είμαστε καλοί δρομής και είχαμε πολλά εμπόδια να ε, υπερβούμε. Και ακόμα και στο τέλος του αγώνα ε, μείναμε, επιμείναμε. Βλέπουμε ότι αλλάζει και το θεσμικό πλαίσιο. Μέσα στη, στα όρια στα νέα όρια της συναπόφασης μπορέσαμε να επιτύχουμε αρκετά. Επιτύχαμε ως προς το θέμα της ευρωπαϊκής διακυβέρνησης και του, του πακέτου των έξι μέτρων. Εάν μιλάμε για καλή οικονομική και πολιτική συνεργασία, φτάσαμε σε μία πολύ καλή συμμαχία στις όχθες του Δούναβη και η Ουγγρική Προεδρία εργάστηκε πολύ σκληρά προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι βεβαίω όλοι ικανοποιημένοι, αλλά νομίζω ότι υπηρετήσαμε όχι μόνο την Ευρώπη, αλλά και την Ουγγαρία και το λαό της. Αρχίζει η διαδικασία Catch the Eye. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω για άλλη μια φορά ότι συνεργαστήκαμε πολύ καλά και με τον Γιάννος Μάλτονη και με την ε, Ενίκο Γκέρι. Και σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, δεσμεύσεις σας και για τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε στο Catch the Eye, Angst για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θερμό ευχαριστώ στην Ουγγρική Προεδρία και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Την κρίνομαι θετικά. Πραγματοποιήθηκε σε εποχή πολλών κρίσεων. Κρίση του ευρώ, πολιτικές κρίσεις στην Αφρική σε σχέση με την άνοιξη των ε, κρατών ή κρίση από το πυρηνικό ατύχημα στην ε, Ιαπωνία. Η Προεδρία επιτυχώς για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και έκανε πολλά πράγματα για την εξέταση των προτύπων ασφαλείας των πυρηνικών εργοστασίων. Σχολήθηκε με δύσκολα θέματα όπως σταθεροποίηση της κρίσης. Δεν μπορώ να ε, συμφωνήσω με τις απόψεις των κυρίων Κονβέντιτ και Φάραντζ που είπαν ότι η Προεδρία αυτή ε, δώσε λύσεις ε, για την κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όμως ευχαριστώ για τις προσπάθειες που κατέβαλε η Ουγγρική Προεδρία. Η κυρία ακούσαμε τον κύριο Όρμπαν να αναφέρεται στην ε, συνεργασία με τα πολιτικά κόμματα. Μίλησε υποτιμητικά. Ε, μετά αναφέρθηκε μόνο στο ΕΛΚ. Υπάρχουν πολλά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όμως έτσι δεν είναι. Όλες οι προεδρίες ε, φραγίστηκαν από κάτι. Εσείς τις ξεπεράσατε όλες ε, με την τροποποίηση του Ουγγρικού Συντάγματος. Ε, ε, αναφέρθηκε από ορισμένους ε, μια άγνοια της Επιτροπής της Βενετίας, ε, άγνοια παράδεκτη. Επίσης αναφέρθηκε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι τόσο σημαντική όσο τα τεκτενόμενα στα κράτη-μέλη. Αυτό δεν είναι καλό παράδειγμα. Μια άλλη προτεραιότητα είναι η βελτίωση της κατάστασης των νέων. Εσείς σε αυτό το τομέα θα ήθελα να ξέρω τι κάνατε, γιατί προσωπικά νομίζω ότι δεν κάνατε τίποτε. Διακοπή ο κύριος Πιετρόφσκι. Ευχαριστώ πολύ. Η Ουγγρική Προεδρία οργανώθηκε σε στιγμή αντιμετώπιση σημαντικών κρίσεων στην Ευρώπη και διεθνώς. Καμία άλλη προεδρεύουσα χώρα δεν μπόρεσε να πετύχει όλους τις τους στόχους. Η Ουγγρική τα κατάφερε πολύ καλά. Πέτυχε την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την Κροατία και την έγκριση του Six Pack. Επίσης κατάφερε να τονιστεί, να δοθεί προσοχή στην περιοχή των παραρδουναβίων περιφερειών και χωρών. Η στρατηγική της Ουγγρικής κυβέρνησης δείχνει πώς είναι ο καλύτερος τρόπος χρησιμοποίησης των ενωσιακών πόρων και η Επίτροπος Ρέντινγκ το τόνισε ότι έκανε προσπάθειες στην Ουγγαρία η Ουγγαρία να προστατευτεί και η ζωή των αγέννητων ακόμη παιδιών. Ο κύριος Όμπερ Μάγερ. Ευχαριστώ πολύ. Η Ουγγρική Προεδρία άρχισε με εσωτερικά πολιτικά γεγονότα που δημιούργησαν ε, ταραχές. Είχαμε την ε, κρίση του ευρώ, τη δημοσιονομική, την αραβική άνοιξη, το ιαπωνικό ατύχημα. Πολλές επιτυχίες σημειώθηκαν, ε, διαπραγματεύσεις με Ισλανδία, ολοκλήρωση διαπραγματεύσεων με την Κροατία, ε, επίσης η στρατηγική για την πυρηνική ενέργεια. Νομίζω ότι εδώ λείπει κάτι όμως και δεν ξέρω αν η διεύρυνση του χώρου Σέγγεν προάγει την ασφάλεια των πολιτών. Γενικά έγινε καλή δουλειά και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους Ούγγρους γείτονες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μίλαν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Όρμπαν, θα ήθελα να σας συγχαρώ εξ ονόματος της σλοβενικής αντιπροσωπείας του ΕΛΚ. Θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Παρά τις δυσχέρειες αναλάβατε μία προεδρία η οποία οποία, η οποία ε, είχε να αντιμετωπίσει ένα πολιτικό ε, τσουνάμι από την ε, αριστερά. Είχατε να αντιμετωπίσετε η Φουκουσίμα, την χρηματοοικονομική κρίση και είχατε να αντιμετωπίσετε και εσωτερικά πολιτικά ζητήματα. Παρά τα πολλαπλά αυτά μέτωπα, αντιμετωπίσατε, τα καταφέρατε αρκετά καλά. Το ευρωπαϊκό εξάμεινο είναι ένας προευρωπαϊκός μηχανισμός ο οποίος εγκρίθηκε μετά από την έγκριση των συνθήκων. Διακόπτει ο πρόεδρος η κυρία Μόνικα Βλασικόβα. Ευχαριστώ πολύ. Η Ουγγρική ε, αντιπροσωπεία ε, πραγματικά αξίζει συγχαρητήρια. Η Προεδρία είχε φιλόδοξο πρόγραμμα και πρέπει να την ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Νομίζω ότι η Ολομέλεια και το Κοινοβούλιο δεν πρέπει να εκφράζουν μόνο κριτική, η χώρα που αναλαμβάνει την Προεδρία επίσης δεν πρέπει να ε, χρησιμοποιεί καταχρηστικά την Προεδρία της. Ε, εσείς κύριε Ορμπάνος, Πρωθυπουργός της χώρας που είχε την Προεδρία, πολύ συχνά κάνατε κατάχρηση της θέσης σας αυτής. Πάντως, πρέπει να σας ευχαριστήσουμε η αρχή όμως ε, δεν ήταν τόσο, η αρχή της Προεδρίας σας δεν ήταν τόσο ευτυχής. Με την ε, παρέμβαση αυτή κλείνει ο κύκλος Catch the Eye. Ζητώ συγγνώμη από εκείνους που δεν ε, μπόρεσαν να παρέμβουν. Καλύψαμε και αυτόν τον γύρο και θα δώσουμε τώρα το λόγο στον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς ο οποίος θα απαντήσει και θα κλείσει τη συζήτηση εξ ονόματος της Επιτροπής. Κύριε Σεύκοβιτς, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητά ε, μέλη, η συζήτηση ε, καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση καθώς και η εκπεριτροπή σε προεδρία. Και το λογότυπο της Ουγγρικής Προεδρίας ήταν για μια δυνατή Ευρώπη. Νομίζω ότι εμπολής ε, ανταποκρίθηκε η Ουγγρική Προεδρία. Ας δούμε την καλύτερη προστασία καταναλωτών, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, το Ρωμά, τη στρατηγική για το Δούναβι, καθώς και οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης της Κροατίας, για να αναφερθούμε σε μερικά ζητήματα, καθώς και η οικονομική διακυβέρνηση. Θα ήθελα επίσης να αντιδράσω στα σχόλια των Ευρωβουλευτών σε σχέση με το Ουγγρικό Σύνταγμα και τη θέση της Επιτροπής επί του θέματος. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και χρειάζεται πολύ προσεκτική ανάλυση πριν φτάσουμε σε συμπεράσματα. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι το νέο Σύνταγμα θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2012 και θα υπάρχουν και εφαρμοστικά μέτρα. Το Σύνταγμα δεν θίγει ζητήματα συμμόρφωσης με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Τα ένομα συμπεράσματα θα ε, ληφθούν υπόψη και θα αποτιμηθούν όταν τεθεί σε εφαρμογή. Επίσης, παρακολουθήσαμε την έκθεση της Βενετίας σε σχέση με τα δεδομένα της 20ης Ιουνίου, καθώς και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αναλύουμε την κατάσταση γι' αυτό μέσα στα πλαίσια του ρόλου μας ως θεματοφύλακα του ευρωπαϊκού δικαίου θα είμαστε, θα επαγρυπνούμε έναντι όλων των κρατών και της Ουγγαρίας και θα χρησιμοποιήσουμε τα προνόμια μας εάν αυτό χρειαστεί. Τώρα, ε, αυτή η Προεδρία, τι επιτέλεσε. Ενισχύσαμε την οικονομική διακυβέρνηση και την ε, κοινή οικονομική πολιτική μέσω της, ε, του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Η τρέχουσα κρίση μας απέστειλε το μήνυμα του πώς βαίνουν οι οικονομίες και πώς το μέλλον μας είναι αλληλένδετο. Μιλάμε για ένα κοινό χώρο των 27 οικονομιών και τι μπορούμε να κάνουμε τη στιγμή που μια χώρα δεν αποδίδει καλώς. Γι' αυτό φτάσαμε στην στρατηγική 2020 και αυτή ήταν και η βάση για το πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ουγγρική Προεδρία για το επιτυχές πρώτο ευρωπαϊκό εξάμεινο και τις ε, ειδικέ συστάσεις τις οποίες ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κάτω από τις καλύτερες δυνατές συνθήκες έτσι ώστε να μεταβούμε από το ευρωπαϊκό στα εθνικά εξάμεινα, διότι οι μεταρρυθμίσεις είναι επιτυχής όταν εφαρμόζονται σωστά από τις εθνικές κυβερνήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο πακέτο οικονομικής διακυβέρνησης και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο επετέλεσαν μεγάλες πρόοδους και νομίζω ότι θα επιτύχουμε ως προς αυτό το πακέτο διακυβέρνησης. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε αυτό το επιπρόσθετο βήμα ως προς τις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα πρέπει, οι οποίες θα πρέπει να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν. Όμως ε, η Ουγγρική Προεδρία τα κατάφερε έτσι ώστε να αποφέρει καρπούς αυτή η πρωτοβουλία. Από την πρώτη ημέρα η Ουγγρική Προεδρία ασχολήθηκε με τη διαπραγμάτευση για την ε, προσχώρηση της Κροατίας. Αυτό ήταν ένα μεγάλο βήμα όχι μόνο για τους Κροάτες αλλά και για όλα τα Δυτικά Βαλκάνια, για τα Δυτικά Βαλκάνια γενικότερα. Πρόκειται για μια αξιόπιστη διαδικασία από πλευράς προετοιμασίας και από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει αναλάβει αυτή την υποχρέωση έναντι των Δυτικών Βαλκανίων. Επίσης διαμορφώθηκαν νέες πολιτικές ως προς ε, την πολιτική γειτονία. Αυτό το επέτυχε η Ουγγρική Προεδρία για τις ε, περιφέρειες αυτές. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημαντικές στρατηγικές. Πρώτον, τη στρατηγική του Δούναβη, όπου θα έχουμε να κάνουμε με μία πρώτη μακροοικονομική στρατηγική μέσα από την κοινή συνεργασία και την πραγματογνωμοσύνη της Κομισιόν μπορούμε να ανορθώσουμε αυτή την περιοχή σε, η οποία θα μετατραπεί σε μια περιοχή ευημερία. Επίσης η στρατηγική υπέρ των Ρωμά ήταν ιδιαίτερα θετική διότι το θέμα των Ρωμά είναι ευρωπαϊκή εμβέλειας θα πρέπει να επιληθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλα τα θεσμικά όργανα, από όλα τα κράτη-μέλη, άρα αυτή η ε, αλληλοεξάρτηση αλληλο, αυτών των ζητημάτων θα οδηγήσει σε θετικά αποτελέσματα για την μειονότητα των Ρωμά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους συνεταίρους μου, τον Υπουργό Εξωτερικών και την Υφυπουργό Γκέρι, οι οποίοι μας συνέδραμαν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεύκοβης και θα τελειώσουμε με αυτό το πολύ σημαντικό θέμα δίνοντας το λόγο στον κύριο Βίκτορ Όρμπαν τον Πρωθυπουργό της ε, ε, Ουγγαρίας. Έχετε το λόγο, κύριε Όρμπαν. Eh, Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Καταρχήν θα ήθελα και πάλι να επαναλάβω ότι η Ουγγρική Προεδρία εκφράζει ε, ευχαριστίες και ευγνωμοσύνη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ολόκληρο το Κοινοβούλιο ναι. εκφράζει ε, επίσης ε, ευχαριστίες στον πρόεδρο Μπούζεκ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μας στήριξε μέχρι το τέλος. Επιτρέψτε μου να επαναλάβω ότι θα ήθελα να εκφράσω ιδιαίτερες ευχαριστίες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τον επικεφαλής του, τον πρόεδρό του για την εξαιρετική πολιτική υποστήριξη. Δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε στερηθεί και να έχουμε τις επιτυχίες που είχαμε χωρίς αυτήν. Από την αρχή η ε, αριστερά μας επετέθη. Αυτό θα μπορούσε να παραλύσει την Προεδρία, θα μπορούσε να μας ε, παρακολύσει από την επίτευξη των στόχων μας. Εμείς έπρεπε να αποκρούσουμε τις επιθέσεις ε, της αριστεράς και χρειάζονταν γι' αυτό η βοήθεια του ΕΛΚ. Είμαι ευγνώμων στο ΕΛΚ που μας παραστάθηκε και μας βοήθησε στο έργο μας. Αξιότιμα μέλη κυρίες και κύριοι, Κάποιες προσωπικές παρατηρήσεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Όχι για προσωπικούς λόγους, αλλά προς το συμφέρον της Ουγγαρίας πρέπει να αποκριθώ. Να αναφερθώ σε ορισμένα θέματα συγκεκριμένα. Νομίζω ότι είναι ευθυνή ρητορία όταν μιλάμε για κακούς ηγέτες και καλούς δημοσίους υπαλλήλους που κάνουν καλά τη δουλειά τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άκουσα πολλές φορές το επιχείρημα αυτό το οποίο πάντα ε, το εκφράζει η αντιπολίτευση όταν αντιμετωπίζει κυβέρνηση η οποία αδιαμφισβήτητα επέτυχε στο έργο της και η αντιπολίτευση δεν θέλει να αναγνωρίσει τα επιτεύγματα των ηγετών αυτών. Ίσως ε, θα ήταν λίγο αστείο επιχείρημα αν δεν γινόταν τόσο κουραστικό λόγω των συχνών επαναλήψεων. Στην Ευρώπη υπάρχουν κυβερνήσεις που επέκριναν και σχολίασαν την Ουγγρική Προεδρία. Δεν αναφέρομαι στις Βρυξέλλες. Δεν υπάρχει ε, Πρωθυπουργό και κυβέρνηση που να δικαιούται να επιβάλλει σύνταγμα στην Ουγγαρία. Μόνο ο ουγγρικός λαός έχει το κυρίαρχο δικαίωμα να αποφασίζει για το σύνταγμά του. Αυτό θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω εδώ. Εμείς ε, πιστεύουμε στις νυφάλιες συζητήσεις στην Ευρώπη και Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απαντήσω στον κύριο Κονμπέντιτ γιατί νομίζω ότι δεν πρόσεξε τη σχετική αναφορά μου. Θα ήθελα λοιπόν να σχολιάσω τις παρατηρήσεις του. Παρακολούθησε το πολιτικό μου έργο και τους λόγους μου στη Βουδαπέστη. Θα ήθελα να επιβεβαιώσω την άποψή μου σύμφωνα με την οποία οι Βρυξέλλες δεν είναι μόσχα. Θα ήθελα αυτό να το καταστήσω όσο γίνεται σαφέστερο. Πάντα θα υπερασπίζομαι την Ουγγαρία απέναντι σε τέτοιες επιθέσεις, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, ακόμα και αν προέρχονται οι επιθέσεις αυτές από τις Βρυξέλλες, διότι δεν θα μας υπαγορεύσετε τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είστε σε θέση να μας το υπαγορεύετε αυτό. Και βεβαίως θα ε, στηρίξω την Ευρώπη αν ε, πω αυτό ακριβώς που λέω, ότι ε, κανείς δεν επιτρέπεται να υπαγορεύσει στην Ουγγαρία τι θα κάνει και τι όχι. Φαίνεται λοιπόν ότι στις πολιτικές μας συζητήσεις και αντιπαραθέσεις ε, πολλοί αναφέρουν ότι υπάρχουν εξεγέρσεις ε, ε εναντίον κάποιων κυβερνήσεων και δικτατοριών. Επίσης ε, αναφέρεται ε, ότι η δημοκρατία λειτουργεί όταν ε, ψηφίζονται ε, οι κυβερνήσεις και όταν βεβαίως τιμωρούνται από την λαϊκή ψήφο. Θα ήθελα να πω ότι εξ ονόματος της Ουγγρικής κυβέρνησης και προσωπικά δεν είμαστε ευρωσκεπτικιστές ε, ούτε σκεπτικοί Δεν είναι στη φύση μας αυτό. Είμαστε ανοιχτοί, πιστεύουμε στα πράγματα, ε, αντιδρούμε ανοιχτά και όχι επιφυλακτικά. Πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, στη συνεργασία. Η... Ανήκω σε μια γενιά, οι παππούδες των οποίων έλεγαν ότι αν δεν υπάρχει ενότητα και συνεργασία στην Ευρώπη, τότε αργά ή γρήγορα θα ξεσπάσει πόλεμο στην Ευρώπη. Εμείς αυτό το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά. Και εμείς ε, είμαστε ε, ένα κράτος, ε, ένα έθνος που υπέφερε από τους δύο παγκοσμίους πολέμους και γι' αυτό είμαστε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ενότητας και Συνεργασίας. Ταυτόχρονα καθιστώ σαφές ότι πάντα θεωρούσα ότι το έργο σας είναι σημαντικό. Ανήκα σε μια κοινότητα στην Ουγγαρία με βασικές αξίες από την Καθολική Εκκλησία. Πάντοτε μια βασική αρχή είναι ότι πρέπει να μεταρρυθμίζουμε την Εκκλησία κάνατε και κάποιες ε, επικριτικές παρατηρήσεις ε, χρήσιμες ε, και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να μεταρρυθμίζουμε την Εκκλησία, άρα κατ' επέκταση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζονται λοιπόν αυτές οι επικριτικές παρατηρήσεις που στηρίζουν το έργο μας προς αυτή την κατεύθυνση. Σε ό,τι αφορά το Σύνταγμα, πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται τις συνταγματικές οντότητες των κρατών μελών. Αυτό είναι κάτι το οποίο προκύπτει σαφώς και αδιαμφισβήτητα απορρέει και από τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς επιμένουμε ότι οι Ούγγροι θα πρέπει να καταρτήσουν και να εγκρίνουν το δικό του σύνταγμα. Ξεκαθαρίζω προς όλους. Ε, όταν μιλάμε για ζωή, οικογένεια, έθνος, όλες αυτές οι αξίες, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, όλα αυτά σφραγίζουν το σύνταγμά μας. Και υποστηρίζονται από εκατομμύρια ανθρώπους. Ο κόσμος χαίρεται όταν ακούει ότι φροντίζουμε για αυτές τις αξίες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχουν μόνο επικριτές της Ουγγαρίας, υπάρχουν άλλοι που ασπάζονται τις αξίες της οικογένειας ε, του έθνους και συμφωνεί με ένα σύνταγμα που αποδίδει αξία σε όλα αυτά. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση που συμφωνούν μαζί μας και θεωρούν ότι το Ουγγρικό Σύνταγμα είναι ένα εξαιρετικό επίτευγμα. Συμπερασματικά, ε, να φροντίσουμε να μην υπάρχουν παρανοήσεις και παρεξηγήσεις μεταξύ μας. Οι αναφορές που έγιναν στην γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας. Θα ήθελα να παραθέσω τρεις φράσεις από την αρχή της γνωμοδότησης. Παραθέτω. Η Ουγγαρία ενέκρινε ένα νέο σύνταγμα το οποίο ανταποκρίνεται τις γενικές ευρωπαϊκές απόψεις σχετικά με το τι είναι αποδεκτό για ένα σύνταγμα. Χαιρετίζω με το γεγονός ότι το Ουγγρικό Σύνταγμα εδράζεται σε τέτοιες βάσεις ώστε να δημιουργεί ε, ένα σύνταγμα συστημάτων που στηρίζει, ε, στηρίζεται στη συνταγματικότητα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Επίσης, το Σύνταγμα ε, συνάδει με τον θεμελιώδη χάρτη ε, ευρωπαϊκών αξιών στην Ευρώπη. Η φύση, η πολιτική φύση του Ουγγρικού Συντάγματος δείχνει ότι είναι ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό σύνταγμα. Οι Ούγγροι και το Ουγγρικό Κοινοβούλιο ε, όπως, προβλέπει, όπως προβλέπουν οι ευρωπαϊκές συνθήκες, θα προχωρήσουν στην έγκριση των εφαρμοστικών τους κανόνων. Θέλω να ευχαριστήσω όσους ε, μας ε, συνεχάρισαν για την Προεδρία μας. Ε, ήταν μεγάλη μου χαρά που συνεργάστηκα μαζί σας τους προηγούμενους μήνες. Ήταν μεγάλη χαρά όχι μόνο να ακούω τους επένους σας, αλλά και να συζητώ μαζί σας. Ξέρω ότι πολλοί ασκήσατε κριτική, γενικά όμως μας αντιμετωπίσατε ε, καλά και θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου προς όλους, συμπεριλαμβανομένης της αριστεράς. Θα ήθελα να σας καλέσω να στηρίξετε την Πολωνική Προεδρία όπως κάνετε και με την Ουγγρική. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πρωθυπουργέ για την παρουσίαση των πεπραγμένων της Ουγγρικής Προεδρίας και για τα σχόλια που μόλις προσθέσατε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Ουγγρική Προεδρία ήταν ιδιαίτερα φιλική προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι εκείνη ενέκρινε τους κανόνες δεοντολογίας για τις σχέσεις μεταξύ Κομισιών Κοινοβουλίου και ως προς τις πολιετής δημοσιονομικές προοπτικές. Αυτό θέλαμε κι εμείς και οι επόμενες προεδρίες θα χρειαστεί να αναλάβουν την ίδια δέσμευση θα ακολουθήσουν δηλαδή το δρόμο που άνοιξε η Ουγγρική Προεδρία και που είναι πολύ θετικός για την επίτευξη των στόχων της πολιετούς αυτής διακυβέρνησης. Σας ευχαριστώ ακόμη μια φορά καθώς και τον Αντιπρόεδρο κύριο Σεύκοβιτς της Επιτροπής και όλους τους συναδέλφους για τη συζήτηση αυτή. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε τη συζήτησή μας, τι συζητήσει μας. Αν τελειώσετε με τα πηγαδάκια αποχαιρετισμών και συγχαρητηρίων, θα συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα, εξίσου σημαντικό. Πρόκειται για την έκθεση της κυρίας